We Λοιπόν, συνεχίζουμε με το σημείο 20 της ημερήσιας διάταξης ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Πρώτη ανακοίνωση ορισμός εισηγητών ε, για γνωμοδοτήσεις η έκθεση για την απόφαση του Συμβουλίου για την εξουδότηση ε, προς τη Ρουμανία να αποδεχθεί την προσχώρηση του Περού στην συνθήκη της Χαϊς του 1980 ανατίθεται στον κύριο Τζαμπάσκι. Δεύτερον, η έκθεση για τις αστικές πτυχές ε, της ε, Διεθνούς Απολογής Παιδιών είχε ανατίθεται επίσης ο κύριο Τζαμπάσκι η έκθεση 4 που αφορά τη συνθήκη της Χάγης για τις αστικές πτυχές ε, συγγνώμη το είπα ήδη το 5 έκθεση για την αναγνώριση δικαιοδοσίας και την εφαρμογή αποφάσεων για ε, γαμικά θέματα ανατίθεται στον κύριο Σβιεύκα και η έκθεση υλοποίησης ε, βάσει της Έκθεση ε, από την Κομισιόν προς το Συμβούλιο για την περιβαλλοντική λογοδοσία όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικών ζημιών ανατίθεται στην κυρία Φεράρα όσον αφορά τις γνωμοδοτήσεις. Uh, uh, ο κατάλογος των τρίτων χωρών, των οποίων οι υπήκοοι πρέπει να διαθέτουν θεωρήσεις κατά την διέλευση των εξωτερικών συνόρων και των χωρών ε, με απαλλαγή ε, ε, όσον αφορά την Ουκρανία πηγαίνει στην κυρία Χάουταλα. Η γνωμοδότηση για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους λόγω έκθεσης καρκινογόνα ή μεταλλαξιογόνα στο χώρο εργασίας, στον κύριο Χρυσόγονο. Οι κανονές και τα πρότυπα ασφαλείας για επιβατικά πλοία στην κυρία Μπερζερό η συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την προστασία ε, των, για την εφαρμογή των ε, νόμων προστασίας των καταναλωτών στον κύριο Χρυσόγωνο. Οι πέντε ζητήματα γεωαποκλεισμού και άλλων μορφών διακριτικής μεταχείρισης ε, βάσει υπηκότητας καταναλωτών αναδειχτές στους σοσιαλιστές δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί όνομα έξι συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών σε σχέση με την πρόληψη, την έρευνα, την, τον εντοπισμό και τη δίωξη ε, ποινικών δικημάτων ανατίθεται στον κύριο Τζαμπάσκι. Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκή, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κυβέρνησης του Καναδά όσον αφορά την εφαρμογή των νόμων ανταγωνισμού τους στον κύριο Λεμπρετόν γενική αναθεώρηση του εσωτερικού κανονισμού του Κοινοβουλίου ανατίθεται σε εμένα συντονισμό ορισμένων διατάξεων που προβλέπονται στην νομοθεσία, στον κανονισμό ή διοικητική δράση στα κράτη-μέλη θα γίνει από το ΕΛΚΑ, δεν υπάρχει ακόμα όνομα. Και τέλο, τελευταία γνωμοδότηση για τι επιλογέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, όσον αφορά τη βελτίωση τη πρόσβαση σε φάρμακα. Ανατίθεται στον κύριο Ντιογόν οι συντονιστές συμφώνησαν να καλέσουν την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συγκριτικής Νομικής Ιστορίας σε μία συνάντηση στο μέλλον και τέλος οι συντονιστές συμφώνησαν να αναθέσουν μια μελέτη στο τμήμα πολιτικής για την ανάλυση της αλληλεπίδρευση της ε, οδηγίας οικολογικού σχεδιασμού και της οδηγίας πώληση ε, σε καταναλωτές. Αυτές είναι οι ανακοινώσεις και συνεχίζουμε με το Όσον αφορά το σημείο 21, η κυρία Χάουταλα είναι η συγγήτρια και ζήτησε αναβολή της ψηφοφορίας για το Σεπτέμβριο. Αναβάλλεται λοιπόν. Σημείο 22 αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοεία. Εκεί θα κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Which one is that? So, no, so it's not it's not electronic. No, this is that's a different one. This is it's this one. In land waterways. Okay. So, amendment 24 has been withdrawn. Λοιπόν, η τροπολογία 24 έχει αποσυρθεί, η τροπολογία 25. Ποιος είναι υπέρ, ποιος είναι κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογίες 26, 27 και 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 29 τώρα. Ναι. Πέρας ψηφοφορία εγκρίνεται. Τροπολογία 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε ξανά. It has been rejected. Απορρίφθηκε. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Παρακαλώ για να είμαστε σίγουροι, ας το τσεκάρουμε άλλη μια φορά. Νομίζω ότι είχε απορριφθεί όμως. ναι, απορρίφθηκε. 32 υπέρ. Κατά. Το ίδιο ας τσεκάρουμε για άλλη μια φορά για να είμαστε βέβαιοι. Yes. <laughs> Uh, rejected. Απορρίπτεται. 33 uh, in favor. υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Οι δύο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3 και 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται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 αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά And it has been rejected. 55 uh, in favor. Ε, απορρίπτεται 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται απορρίπτε συγγνώμη 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 και 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 και 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά να τσεκάρουμε ηλεκτρονικά Okay. Adopted. Εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και ψηφίζουμε του συνόλου της του κειμένου, άρχεται η ψηφοφορία. That Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια λοιπόν στην κυρία Μπερζέρο. Then uh, we vote on... Τώρα θα ψηφίσουμε το σημείο 23. Προστασία από τις συνέπειες της εξοεδαφικής εφαρμογής ορισμένων νόμων Ποιο είναι αυτό, λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην κυρία Φεράρα. Και αυτό ήταν. Αυτές ήταν οι ψηφοφορίες. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με το σημείο 24. Ακρόαση. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε με μία ακρόαση για τις προθεσμίες παραγραφής όσον αφορά τα τροχαία ατυχήματα, η σημερινή κατάσταση και τα επόμενα βήματα. Παρακαλώ να κάνετε ησυχία. Thank you very uh, Uh, λοιπόν, ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση στους αξιότιμους ομιλητές. Δυστυχώς είναι κάτι που δεν μπορούσαμε να αποφύγουμε. Και γι' αυτό να πω ότι ξεκινούμε λέγοντας με, ότι είναι μεγάλη μας χαρά που βρίσκονται εδώ μαζί μας οι αξιότιμοι ομιλητές είναι μια κρόση που οργανώνει η Επιτροπή μας. Είναι πολύ ενδιαφέρον για μένα προσωπικά διότι είμαι και εισηγητής για αυτό το θέμα και πραγματικά θα ακούσω με μεγάλη ενδιαφέρον αυτά που θέλετε να πείτε. Οι προθεσμίες παραγραφής ε, για τις αξιόπινες ε, πράξεις διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών. Στην υπηρετική Ευρώπη υπάρχουν ε, διαδικασίες παραγραφής αποσβεστικής, δηλαδή αποσβαίνεται η αξίωση μετά από αυτή την προθεσμία, ενώ σε άλλες χώρες υπάρχουν μόνο περίοδοι παραγραφής βάση της οποίας το δικαίωμα αξίωσης παραγράφεται, αλλά όχι η αξίωση αυτή καθεαυτή. Αυτές οι διαφορές στα εθνικά δίκαια υπάρχουν και ως προς την έναρξη της χρονικής περίοδου Ειδικά για τους ανήλικους και του άτομα με αναπηρία υπάρχει κάποια διάκριση και υπάρχει και διαφορά ως προς το δικαίωμα διακοπής αυτής της περίοδου. Ε, ε, επειδή υπάρχει διαφορά ως προς το διάστημα έναρξης της διαδικασίας. Υπάρχει επίσης διαφορά ως προς ε, το κράτος ε, ε, στο οποίο έγινε το ατύχημα. Η εθνική νομοθεσία λοιπόν πρέπει να, ε, να ομολογήσουμε ότι είναι ιδιαίτερα σύνθετη και τα θύματα, οι ζημιοθέτες δεν γνωρίζουν τους κανόνες των κρατών μελών στα οποία ταξιδεύουν. Αυτό σε συνδυασμό με τις διαφορές στην νομοθεσία για την παραγραφή μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες ε, συνέπειες για τα θύματα ε, που δεν θα μπορέσουν να καταθέσουν ε, ενδεχομένως εγκαίρως την αξίωσή τους, την προσφυγή τους, αλλά και να αποζημιωθούν σωστά ή θα πρέπει να καταβάλουν πολλές δαπάνες δικαστικές. Έχουμε τώρα την έκθεση του Dr. Μάρκο Μπόνα και της Τζένι Παπέτας που ε, είναι οι άνθρωποι στους οποίους ε, δόθηκε ε, η εντολή να κάνουν μια έκθεση για την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για το θέμα αυτό. Σήμερα έχουμε μια ηχογραφημένη και μάλλον μαγνητοσκοπημένη παρουσίαση και μια επεξήγηση του λόγου που ξεκίνησε αυτή η αξιολόγηση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Εμείς θέλουμε τα μέλη του Κοινοβουλίου, οι ειδικοί και οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να συζητήσουν για τη σύγκληση σχετικά με τις περιόδους παραγραφής για τα διασυνοριακά τροχαία ατυχήματα. Οι εκπρόσωποι από ευρωπαϊκές οργανώσεις ε, ε, δικηγόρων για προσωπική βλάβη, από ασφαλιστικές εταιρείες, από θύματα τροχαίων κτλ. θα συνεισφέρουν σε αυτή τη συζήτηση. Πριν δώσω το λόγο στον πρώτο μιλητή για σήμερα, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι υπάρχει ε, στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή live η συνεδρίασή μας και θα καταγραφεί επίσης, θα μηχανητοσκοπηθεί η συνεδρίαση και η ακρόαση. Τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Φίλιπ Μιτ, μέλος του Γενικού Συμβουλίου για την Αγγλία και την Ουαλία και της Ακαδημαϊκής Επιτροπής της Πανευρωπαϊκής Οργάνωσης ε, Δικηγόρων για ε, προσωπικής, ε, προσωπικού ενδιαφέροντος. Αυτός ο οργανισμός, το POPIL, έχει ενεργά δράσει σε αυτό τον τομέα, έχει εκδώσει πολλά ε, πολλές εργασίες ε, για τα τροχαία ατυχήματα και τις περιόδους ε, απαραγραφής. Ο κύριος Σμίτ πρέπει να ξέρει ότι πρέπει να μιλήσει μόνο 10 λεπτά εξαιτία της καθυστέρησης που είχαμε. Ευχαριστώ. Um, um, Καλημέρα. Μετά τα γεγονότα της 23ης Ιουνίου, ε, δεν θα θέσω την ε, άποψη της Βρετανίας, την οπτική γωνία ας πούμε, γιατί ε, έχουμε και το διαταραχή του μετατραυματικού στρες από τροχαία ατυχήματα, αλλά τώρα εγώ πάσχω από μετατραυματική διαταραχή λόγω του Brexit. Η θέση μου λοιπόν εδώ σήμερα είναι ως μέλος της Ευρωπαϊκής πανευρωπαϊκής αυτής ομοσπονδίας που εκπροσωπώ. Δεν εκπροσωπώ λοιπόν τη Βρετανική οπτική γωνία, αλλά την άποψη όλων των δικηγόρων που ασκούν τα καθήκοντά τους σε αυτό το τομέα και ειδικεύονται στις ε, αξιώσεις για τροχιά ατυχήματα. Έχω προετοιμάσει μια εργασία ε, την οποία μπορείτε να δείτε ε, είναι διαθέσιμη. Θα μιλήσω για 10 λεπτά. Το πλαίσιο είναι πολύ σημαντικό. Να σας ε, θυμίσω ε, ποιο είναι η νομοθετική πρόοδος που έχει επιτευχθεί ως τώρα. Έχουμε την κωδικοποιητική οδηγία 2009 103 ΕΚ που εναρμονίζει τα ελάχιστα, τις ελάχιστες προδιαγραφές για την παροχή ασφάλιση μη ζωή και την κατάργηση των ελέγχων για την ασφαλιστική κάλυψη. Να πω ότι αυτό που φαίνεται είναι ότι πρέπει να αναπτύξουμε τη σημαντική αρχή της παροχής συγκρίσιμης αντιμετώπισης για τα θύματα των τροχαίων ατυχημάτων, ανεξάρτητα από το ατύχημα. Ε, ήδη έχουμε την παροχή ελάχιστης κάλυψης Δηλαδή γίνεται πλήρης αποζημίωση και λογική και δίκαιη των θυμάτων. Επίσης ε, υπάρχει ε, το δικαίωμα ευθείας αγωγής που είναι ευρωπαϊκό και όχι εθνικό και έχουμε και το δικαίωμα κοινοποίηση μιας αξίωσης σε έναν διεκπαιρεωτή στη χώρα ε, του ενάγοντος ε, χρησιμοποιώντας τις διαδικασίες που γνωρίζει ο ενάγον. Αυτά είναι τα στοιχεία που κατά την άποψή μου πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ως βάση. Έχουμε λοιπόν επίσης την εξαγωγή ενός συστήματος διακανονισμού των αξιώσεων στη χώρα ε, όπου ζει ο ενάγων και έχουμε και την ε, παροχή του δικαιώματος ε, προσφυγής έναντι του ασφαλιστή. Ε, αυτό το δικαίωμα ε, είναι στη χώρα που ζει ο ζημιωθής. Όμως ε, το ίδιο δίκαιο που υφίσταται και εφαρμόζεται για μια τέτοια αξίωση γίνεται με αναφορά στο δίκαιο περί αδικοπραξιών που ισχύει στη χώρα αυτή. Το οποίο δίκαιο είναι αυτό είτε της χώρας όπου έλαβε χώρα το τροχαίο, είτε αυτό στο οποίο συνήφθη ε, το ασφαλιστικό συμβόλαιο σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού. Έχουμε αυτή λοιπόν τη διαφορά. Από τη μία την κωδικοποιητική οδηγία η οποία ως βασικό στόχο έχει τα προδιαγραφές για τη δίκαιη πρόσβαση στη δικαιοσύνη των θυμάτων και τις διαδικασίες που θα επιτρέπουν τους ενάγοντες να διακανονίζουν μια αξίωση στη χώρα τους που γνωρίζουν το σύστημα και υπάρχει και το ε, θέμα της νομικής διαδικασίας που ε, συνήθως ε, έχει να κάνει με το δίκαιο της χώρας στην οποία έγινε το ατύχημα, συχνά ξένο δίκαιο και αυτό αποκλείει τους ενάγοντες ή τους δικηγόρους από τη γνώση. Εμείς θεωρούμε ότι εδώ υπάρχει φραγμό στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη γιατί υπάρχει διαφοροποίηση και αβεβαιότητα σε σχέση με την εφαρμογή των κανόνων, ποιοι κανόνες ισχύουν. Έτσι κάποιες αξιώσεις δεν ε, διώκονται είτε επειδή δεν υπάρχει χρόνος, έχει παρέλθει η προθεσμία παραγραφής ή επειδή αυτό θεωρείται ότι ισχύει. Γιατί οι δικηγόροι στη χώρα του ενάγοντος δεν κατανοούν ε, το σύστημα σε άλλες δικαιοδοσίες. Και οι δυσκολίες προκύπτουν από το γεγονός της διαφοράς της περίοδου παραγραφής ένα έτος στην Ισπανία, 10 στη Γαλλία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορείς να ε, κάνεις επέκταση αυτής της προθεσμία σε άλλες χώρες όχι. Επίσης ξεκινά διαφορετικά να τρέχει αυτή η προθεσμία ε, σε κάποιες χώρες ε, μπορεί να υπάρχουν παιδιά, ας πούμε, ή ασθενείς άτομα χωρίς τη δυνατότητα να δράσουν για τον εαυτό τους, έχουν διαφορετική ε, αντιμετώπιση. Σε κάποιες άλλες χώρες η ποινική διαδικασία σταματά το ρολόγι, σε άλλες χώρες μπορεί να διακοπεί η, η περίοδος αυτή για κάποιο διάστημα, σε άλλες όχι. Είτε με επίδοση είτε με έκδοση απόφαση είτε με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία. Ε, το γεγονός ότι υπάρχει λοιπόν μια σύνθετη εικόνα οδηγεί σε ε, διακρίσεις έναντι των ευάλωτων ομάδων όπως είναι τα παιδιά και οι άνθρωποι που είναι ανίκανοι ε, για να εκπροσωπήσουν τον εαυτό τους. Επίσης, να πω ότι σχετικά με τα παιδιά τα παιδιά έχουν μεγαλύτερη πρόσταση, ας πούμε, στο Ηνωμένο Βασίλειο από τις άλλες ε, δικαιοδοσίες και υπάρχει κίνδυνος να χάσουν αυτές οι συγκεκριμένες κατηγορίες. Επίσης έχουμε δορυφορικές διαδικασίες, δηλαδή το δίκαιο της ε, χώρας όπου έγινε το τροχαίο ε, είναι πρόβλημα γιατί υπάρχει παραγραφή που δεν θα υπήρχε στη χώρα του ανάγοντος. Επίσης οι δικηγόροι πάντοτε πρέπει να διασφαλίσουν ότι δεν θα έχουν ε, ότι θα πάρουν κάποιε περαιτέρω συμβουλέ από ντόπιου δικηγόρου σχετικά με τι παραγραφέ, άρα έχουμε επιπλέον ε, και γι' αυτό πολλέ φορέ συγκεντρώνουν μαζί πολλού ε, ε κατηγορούμενου ε, για να έχουν εξοικονόμηση. Επίση, υπάρχουν κάποιοι δικηγόροι που δεν αναλαμβάνουν τις υποθέσεις επειδή θεωρούν ότι έχει παραγραφεί η υπόθεση και δεν καταλαβαίνουν ποιες δυνατότητες έχουν να συνεχίσουν. Ε, άρα αυτή η πολυπλοκότητα στην ουσία αποτρέπει ε, από την απονομή δικαιοσύνη. Ε, δεν δίνει κανείς μια μάχη που θεωρεί ότι θα χάσει και αυτό είναι μειονέκτημα, είναι διάκριση. Επίσης, θεωρώ ότι υπάρχει υπάρχουν κανόνες παραγραφής, διότι αυτή είναι η δημόσια πολιτική. Δεν πρέπει από μια συγκεκριμένη περίοδο και μετά να ε, διώκεται κάποιος, ακόμα και αν υφίσταται η αξίωση. Ποια είναι εκείνη η πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε το υποχρεωτικό ε, δικαίωμα ευθεία αγωγής έναντι των ασφαλιστών, όμως υπάρχει και η ευρωπαϊκή πολιτική που το διευκολύνει αυτό σύμφωνα με το, ε, που ανατρέπει με αναφορά στο εθνικό δίκαιο. Έχουμε την ε, οδηγία για την ευθύνη των προϊόντων που ρυθμίζει ακριβώς ε, την παραγραφή για αξιώσεις για προσωπική βλάβη. Υπάρχει λοιπόν το προηγούμενο, αλλά υπάρχουν και ανομαλίες. Η κωδικοποιητική οδηγία αφήνει το δικαίωμα της πρόσβασης της δικαιοσύνης σε όλους, αλλά αφήνει εκτεθειμένα τα παιδιά και τα άτομα σε αδυναμία εκπροσώπησης. Ε, οι ανομαλίες ε, που αναφέραμε εδώ έχουν ως εξής. Γιατί οι ε, ασφαλιστές και ασφαλιζόμενοι της αλφα να μην μπορούν να ε, έχουν ε, προστασία για ένα θύμα που είναι στη β' αγορά γιατί η πολιτική ενός άλλου κράτους μέλος, ας πούμε της αγοράς β' ε, που επιτρέπει να καλύπτονται αυτοί οι κίνδυνοι στη χώρα δεν μπορεί να καλύψει αυτούς της αγοράς α γιατί οι ασφαλιστές στην αγορά α να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ενώ τα θύματα μειονέκτημα. Η λειτουργία λοιπόν της ενιαίας αγοράς για την ασφάλεια μη ζωής διευκολύνει ε, να έχουμε ασφάλιση μεταξύ των διαφόρων αγορών γιατί οι ασφαλιστές στην αγορά Α και Β όταν είναι η ίδια εταιρεία εποφελούνται από διαφορετικές συνθήκες όταν έχουμε την ενιαία αγορά. Από την άποψη λοιπόν της ενιαίας αγοράς υπάρχουν ανομαλίες ως προς τον δίκαιο ανταγωνισμό, όπως υπάρχουν ανομαλίες και σε σχέση με την προστασία των θυμάτων ε, για το θέμα της παραγραφής. Άρα, ε, θεωρούμε ότι δεδομένου ότι υπάρχει το δικαίωμα ευθείας αγωγής σε σχέση με τα θύματα, οι ανομαλίες αυτές θα πρέπει να εναρμονιστούν με προστασία μέσω του, ε, της εναρμόνισης ε, του δικαίου που αφορά στην παραγραφή. Ε, ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς για όλα αυτά που μας είπατε. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των ασφαλιστών και την άποψη των ε, θυμάτων, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Νίκολα Ζων Μαρ, ο οποίος είναι επικεφαλής ε, ε, για θέματα μικροοικονομικά τον οργανισμό στον οποίο εργάζεται και θα μας παρουσιάσει την ομιλία του με τον κύριο Κίον Φαν ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος της ε, Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ε, των ε, θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων. Κάθε ένας από εσά, αν έχει την καλοσύνη, 10 λεπτά και λυπάμαι πάρα πολύ που δεν προέφερα και σωστά τα ονόματά σας. Πρώτα απ' όλα δίνω το λόγο στον κύριο Ζαν σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σβόμποντα. Σας ευχαριστώ που μας δώσατε τη δυνατότητα να συμμετέχουμε σε αυτή την ακρόαση για τις ε, περιόδους παραγραφής. Η δική μου η Ένωση Trans Europe είναι μία ομοσπονδία η οποία εκπροσωπεί 34 μέλη ε, και εκπροσωπούμε περίπου το 95% των ε, εσόδων ε, ασφαλίστρων για αυτόν τον τομέα. Εμείς εκπροσωπούμε περίπου το 1 τρίτο ε, των ασφαλίστρων εκτός ασφάλειας ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. αλλά δηλαδή μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να συμμετάσχουμε σε οποιαδήποτε συζήτηση ε, αφορά τα δικά μας τα συμφέροντα. Ο στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι τα θύματα από τροχιά ατυχήματα προστατεύονται παρκώς και γι' αυτό το λόγο χαιρετίζουμε και εμείς τη δυνατότητα που μας προσφέρεται να συμμετάσχουμε στη συζήτηση. Ε, θα ήθελα να πω πρώτα απ' όλα κάποια λόγια για την, το το δικό μας το ρόλο στην ε, προστασία των τιμάτων και το τι ακριβώς ισχύει και μετά θα περάσω στο θέμα πιο συγκεκριμένα των περίοδων παραγραφής σε σχέση με το πρόβλημα και σε σχέση με ενδεχόμενες λύσεις. Και εδώ θα δείξω και το θέμα της ενημέρωσης και της εναρμόνισης. Ξεκινάω λοιπόν με κάποια λόγια για το ενωσιακό πλαίσιο και πού ακριβώ λειτουργεί η Motor Insurance. Η δική μας οδηγία, η οδηγία που μας αφορά, έχει ως βασικό στόχο να διασφαλίσουμε ότι τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων ε, σε όλη την ενωσιακή επικράτεια. Υπάρχει λοιπόν μια σειρά σημαντικών διατάξεων για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος και περιλαμβάνονται στην σχετική κωδικοποιημένη οδηγία η οποία ανάγεται στο 2009. Δύο άλλοι βασικοί στόχοι της οδηγίας, ε, που έχει σχέση βέβαια με την πρώτη, είναι να διευκολύνεται η ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασική διάταξη αυτής της οδηγίας λέει ότι θα πρέπει όλα τα <clears throat> οχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να καλύπτονται από ασφάλεια ευθύνης. Εμείς ε, φροντίσαμε να συμπεριληφθούν και κάποιες διατάξεις ε, που προβλέπουν αποζημίωση για την περίπτωση θυμάτων και πώς πιο εύκολα μπορούν τα θύματα να έχουν πρόσβαση σε τέτοιου είδους αποζημίωση. Δηλαδή, οι διατάξεις περιλαμβάνουν το ότι να υπάρχουν εθνικοί οργανισμοί οι οποίοι ε, θα μπορούν να διαπιστώνουν κατά πόσον ο υπάρχει ασφάλεια ή όχι των άμεσα ενδιαφερομένων. Η απάντηση να είναι μέσα σε τρεις μήνες από την ώρα που κατατίθεται η αγωγή αποζημίωσης και επίσης η οδηγία διασφαλίζει ότι τα θύματα έχουν δικαίωμα να αξιώσουν, να υποβάλουν αξίωση στο δικό τους το κράτος μέλος και όχι εκεί που έλαβε χώρα το τροχαίο ατύχημα. Αυτή λοιπόν ήταν μια σύντομη εισαγωγή και θέλω να σας πω ότι κατά την άποψή μας το σύστημα αποζημίωσης που ισχύει είναι ικανοποιητικό για τα ε, θύματα τροχαίων ατυχημάτων, άρα πρέπει να διατηρηθεί. Τώρα, η προοπτική της Trans Europe όσον αφορά τις περιόδους παραγραφής ε, για τροχαία ατυχήματα. Αυτό το θέμα το εξετάσαμε όταν συζητήθηκε μετά από πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 7 και το 8 και η Κομισιόν διεξήγαγε διαβουλεύσεις το 2009 και το 2012. Τα σχόλιά μου βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις συζητήσεις που είχαμε με όλα τα μέλη και τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Τα μέλη τα δικά μας έχουν άποψη που παραμένει ε, αμετάβλητη. Βεβαίως ευχαρίστω να συζητήσουμε και άλλα θέματα που ενδεχομένως να προκύψουν μετά από μελέτη που διεξήγαγαν οι υπηρεσίες στο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα παρουσιαστούν αργότερα. Το ερώτημα που τίθεται σήμερα στην ακρόαση είναι κατά πόσον υπάρχουν ίσως ειδικέ δυσκολίε για τα θύματα τροχιών ατυχημάτων και αυτό ως αποτέλεσμα του ότι υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες παραγραφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς ακριβώς μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτέ οι δυσκολίε. Οι δυσκολίε ε, αντιμετωπίζονται ότι εντάσσονται σε δύο διαφορετικές κατηγορίες. Υπάρχουν περίοδες παραγραφή σε σωσμένα κράτη-μέλη που κρίνονται πολύ ε, για να κατατεθούν αγωγέ ή ε, δεν υπάρχει η σωστή ενημέρωση ε, στα κράτη-μέλη. Το πρώτο ερώτημα που τίθεται είναι πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή τα θύματα τέτοιων ατυχημάτων πόσες φορές χρησιμοποιούν δυσκολίες ακριβώς λόγω του ότι είναι βραχίδιες αυτές οι διατάξεις. Ε, το πιο σημαντικό είναι να γίνει το πρώτο βήμα. Έτσι θα εξευρεθεί η λύση. Και με βάση τις πληροφορίες που έχουμε, το πρόβλημα είναι αρκετά περιορισμένο η μελέτη της Κομισιόν του 2009 αναφέρει ότι υπάρχουν ε, περιπτώσεις δικαστηρίων που έχουν απορρίψει η σχετική αγωγή λόγω του ότι έχει παραγραφεί το αδίκημα, αλλά αυτές οι περιπτώσεις πρέπει να σας πω είναι αρκετά περιορισμένες και εκεί καταλήγει η μελέτη. Για να το κατανοήσει κανείς αυτό πρέπει να έχει κατά νου ότι πρακτικά μόνο ένα μικρό ποσοστό των τροχιών τυχημάτων είναι διασυνεωριακά. Τα περισσότερα θύματα τροχαίων ατυχημάτων, ε, καταπέμπουν σε νομικές συμβουλές ε, και ως εκ τούτου ο νομικός σύμβουλος θα ε, θίξει και θα τοποθετήσει το όλο θέμα. Επίσης γίνονται πολύ φιλικοί διακανονισμοί εκτός δικαστηρίων και κάτι άλλο στις λίγες περιπτώσεις όπου εκπνέει περίοδος παραγραφής προκύπτει κάποιος φιλικός διακανονισμός. Ο αριθμός των θυμάτων που θίγεται, σας είπα και πριν, είναι αρκετά περιορισμένος. Άρα δηλαδή η καλύτερη λύση θα ήταν εκείνη που θα οδηγούσε στο να μην υπερκεραστεί το πλαίσιο που υπάρχει Εκεί κατέληξε η Κομισιόν μετά από τις διαβουλεύσεις του 2012. Άρα δηλαδή ποιες είναι οι λύσεις που προτείνουμε. Στις διαβουλεύσεις του 2012 ε, εξετάσαμε δύο δυνατότητες λύσεων ως Κομισιόν είτε να δίδονται πληροφορίες για τις διαφορές που υπάρχουν στις περιόδους παραγραφής ή να εναρμονιστούν κάποια στοιχεία των κανονισμών για την παραγραφή όταν πρόκειται πιο συγκεκριμένα για διασυνοριακό τροχαίο ατύχημα. Κατά την άποψή μας το να προσφέρονται σωστές πληροφορίες αυτό είναι το καλύτερο και η Insurance Europe ε, δεν ήταν μόνη τη, Τότε και η Κομισιόν διαπίστωσε ότι οι πληροφορίες για τις περιόδους ε, παραγραφής ε, ε, πράγματι αυτό το στηρίζουν όλοι. Και τότε είχαμε πει ότι η ενημέρωση για διαφορετικές περιόδους παραγραφής στα κράτη-μέλη, αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο πόρταλ της Κομισιόν EU Justice σε όλες τις γλώσσες για να υπάρχει σιγουριά ότι όλα τα θύματα θα ενημερώνονται με τον ίδιο τρόπο. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι γενικές αλλά και αρκετά ειδικέ για να καλύπτουν τις ε, ανάγκες. Έτσι λοιπόν θεωρούμε ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο δυσκολιών λόγω των διαφορετικών περίοδων παραγραφής και είναι και ο καλύτερος τρόπος για να στηριχθούν τα θύματα των διασυνοριακών ατυχημάτων. Η άλλη λύση που εξέτασε η Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν η εναρμόνιση των ε, περιόδων παραγραφής για διασυνοριακά ατυχήματα. Κατά την άποψή μας ε, ε, αυτό δεν ξέρουμε αν είναι ικανοποιητικό και πρέπει κανείς να δει και πόσο εύκολο είναι πρακτικά να εναρμονιστούν οι κανόνες. Η απάντηση είναι ότι όλα αυτά είναι πολύ περίπλοκα. Όχι διότι οι νόμοι για τις περιόδους παραγραφής σχετίζονται και με άλλους παράγοντες όπως το είδος των αγωγών που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο, τα αποδεικτικά στοιχεία για να τεκμηριωθεί μια αγωγή και ε, όλοι οι άλλοι περιορισμοί που ενδεχομένω να υφίστανται. Αυτά επηρεάζουν όχι μόνο τη διάρκεια της περίοδου παραγραφής, αλλά και όλους τους άλλους κανόνες που έχουν σχέση με την κατάθεση, την αναστολή και την ε, ε, πάυση αυτής της αγωγής. Επίσης, όλα αυτά μπορούν να επηρεάζουν και την περίοδο παραγραφής. Έτσι λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι το να τροποποιηθούν οι κανόνες αυτό είναι αναπόφευκτο, αλλά αυτό σημαίνει όμως ότι παρεμβαλόμεθα στις εθνικές αρμοδιότητες. Πρέπει να έχουμε κατά νου. Οι διαφορές στις περιόδους παραγραφής αφορούν μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό των διασυνοριακών ατυχημάτων. Γι' αυτό κλείνω λέγοντας ότι δεν αξίζει τον κόπο και γι' αυτό το λόγο ευχαριστώ και άλλη μια φορά το Κοινοβούλιο για αυτά που μας είπε, που μας κάλεσε που μας κάλεσε για να επιβεβαιώσουμε ότι μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα όλο αυτό το θέμα, κυρίως γιατί σήμερα ειδικά πρόκειται να δημοσιοποιηθεί η σχετική μελέτη. Και τώρα το λόγο έχει ο κ. Φανφοντεκέμε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. είναι δύσκολο να προφέρετε το όνομά μου, το έχω συνηθίσει γιατί και οι Ολλανδοί, οι συμπατριώτες μου δυσκολεύονται. Θα είμαι πολύ σύντομο όμως και για να είμαι σύντομο, θα τα πω και στα γαλλικά. Να πω ότι είμαι εκτελεστικό διευθυντή της Ένωσης Γονέων των Παιδιών τα Τροχαίων που είναι βελγική οργάνωση και είναι και μέλος ε, της Ομοσπονδίας της Ευρωπαϊκής ε, FBVR. Εκεί είμαι και μέλος ε, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Για να διευκολύνω τη ζωή μου θα τα συνεχίσω όμως τα γαλλικά. Η Ομοσπονδία λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Θυμάτων Τροχαίων, ΕΒΕΡ... Δεν έχουμε ακόμη ούτε συντομογραφία, ούτε ονομασία στα αγγλικά. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την Νομική Επιτροπή που μας κάλεσε να συμμετέχουμε σε αυτή την ε, ακροασία, την παραγραφή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιστεύουμε, να μπει η διάσταση των θυμάτων ε, στη συζήτηση αυτή και σίγουρα ε, ιδίως όταν μιλάμε για ε, ζητήματα διαγραφής. Και βέβαια για να σας δώσω Έχουμε 25 χρόνια ε, ζωή στην Ομοσπονδία μας. Ε, έχουμε μέλη 25 εθνικές περιφερειακές οργανώσεις. από 17 χώρε. Δηλαδή κάποιε φορές περισσότερες τη μια οργανώση από μια χώρα και η αποστολή μα μεταξύ άλλων είναι η παροχή υποστήριξη των θυμάτων των τραχαίων όλες τι κατηγορίες, όχι μόνο οικογένειε που πενθούν το χαμό ενός παιδιού ή ενός άλλου αγαπημένου προσώπου τη οικογένεια. αλλά και τραυματίες, και τις δικές τους οικογένειες. Ε, στηρίζουμε και ψυχολογικά και βέβαια και τον προσανατολισμό του στη συνδρομή που τους παρέχουμε σε περίπτωση νομικής διαδικασίας κτλ. Όπως επίσης ευαισθητοποίηση και πέδευση για την οδική ασφάλεια. κάτι πολύ ε, θετικό. Έτσι το αντιλαμβάνονται οι συγγενείς ε, των θυμάτων ε, στο δράμα αυτό το οποίο ζουν. Συμμετέχουμε επίσης σε διάφορες άλλες οργανώσεις, ETSC, την Παγκόσμια Συμμαχία, ΜΣΕΕ και άλλες. Έχουμε επίσης ε, ε, πρωτοστατήσει στην ανακήρυξη το 2005 μια ημέρα μνήμης για τα θύματα τροχαίων. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε μια καλή προσέγγιση και ενώπιον δημόσιων φορέων και σε ευτικό επίπεδο για μια καλύτερη προσέγγιση μετά το τροχαίο, δηλαδή υποστήριξη των θυμάτων, των τραυματιών, ε, τη στη δυνατή ιατρική περίθαλψη, δυναμική συνδρομή, όσο μπορούμε να μειώσουμε, να απαλύνουμε τον αντίκτυπο του τροχαίου και να προωθήσουμε την αποκατάσταση ευρυτέρα τι ενία Επίσης ε, σήμερα δεν είμαστε εδώ πιο πολύ για τεχνικούς νομικούς λόγους αλλά για να ε, σας παρακαλέσουμε να συμπεριλάβετε μια διαδικασία, μια προσέγγιση ενσυναίσθηση στις και αποφάσεις που λαμβάνεται σε επίπεδο παραγραφής και προθεσμίας και νομίζω ότι ήδη στην ακρόαση φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η προσέγγιση, αυτή η ενσυναίσθηση. Να πω δύο-τρία πράγματα για τη φάση της ε, αποκατάστασης ε, της βλάβης που ε, φύστανται τα θύματα τροχαίων η διαδικασία και για τα θύματα και για τους συγγενείς τους είναι μια πολύ οδυνηρή εμπειρία. Πολλές φορές οδηγεί σε κάτι το οποίο ζούμε μια δευτερεογενή θυματοποίηση, η οποία μπορεί να ε, πραγματοποιηθεί σε διάφορες ε, φάσεις. Ε, το timing επίσης πάνω απ' όλα είναι κάτι πολύ λεπτό, πολύ ευαίσθητο και η παραγραφή είναι κάτι που εντάσσεται σε αυτή την όλη κατάσταση. Δεν θα πρέπει να γίνουν τα πράγματα ούτε πολύ γρήγορα ούτε πολύ αργά αλλά την κατάλληλη στιγμή. Και αυτό ακριβώς το υποστηρίζουμε και οι επιθεωρητές των ασφαλιστικών εταιρών κτλ. Ε, είναι ένα θέμα να δούμε πότε θα προσεγγίσουμε το θέμα την οικογένεια ενός ε, θύματος, ενός νεκρού, για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία αποκατάστασης. Η διεκδίκηση αποζημίωση μετά το χαμένο ανθρώπου δεν είναι κάτι που είναι το πρώτο πράγμα που έχετε στο μυαλό ε, των ανθρώπων που έχουν χάσει ένα δικό τους. Δεν έχουν το μυαλό για κάτι τέτοιο θα έλεγα. Ε, η κατάλληλη στιγμή, αν θέλετε, είναι μια αποστολή, ένα ειδικό καθήκον για τους ασφαλιστές. Εμείς ε, και τα μέλη μας ε, διαπιστώνουμε ότι η παραγραφή τελικά είναι, δημιουργεί πολύ λιγότερα προβλήματα, δηλαδή είναι σπάνιο. Θα δούμε σε ποιες χώρες έχουν την έδρα αυτές οι οργανώσεις που το λένε αυτά, αλλά τέλος πάντων. Πιο πολλά προβλήματα δημιουργεί το μάκρος των ε, διαπραγματεύσεων των δικαστικών ή των δικών. Διότι εκεί ε, πολλές φορές δημιουργείται απογοήτευση και όπως είπα και η δευτερογενή θυματοποίηση ή η δυσαρέσκεια ε, που νιώθουν τα άτομα τα οποία θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί. Οι επιθεωρητές, διαχειριστές ε, των φακέλων, οι ασφαλιστικές δηλαδή εταιρείε, αλλά και οι δικαστές, δικηγόροι, οι πραγματογνώμονες λοιπά έχουν μεγάλη ευθύνη και πρέπει να διαπιστώσουμε δυστυχώς ότι μέσα σε 20 χρόνια περίπου θα έλεγα δεν έχουν αλλάξει και πολύ τα πράγματα πόσο μάλλον ε, να, έχουν βελτιωθεί αλλά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Πρέπει να ξέρετε επίσης ότι ο η δικαστική πτυχή, ε, το δικαστικό σκέλος ενός τροχιού συχνά συνιστά την πρώτη, εντελώς πρώτη επαφή της οικογένειας του θύματος με το δίκαιο, με το δικαστήριο, με τη δίκη, μια ποινική διαδικασία, αστική διαδικασία. Άρα νομίζω ότι πρέπει να πούμε ε, κάποια πράγματα σε σχέση με την έννοια της αποσβεστικής παραγραφής είναι αποδεκτή αυτή η έννοια νομπονομικής πλευράς. Είναι σημαντικό οι θυγόμενοι να γνωρίζουν ε, τι είναι αυτό ακριβώς, τι θα πει αποκατάσταση της ε, βλάβης που έχουν υποστεί. Και γι' αυτό πρέπει να τα εξηγούμε τα πράγματα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τι θα πει αυτό μετά το τροχαίο, οι δημόσιε αρχέ, δηλαδή πρώτα απ' όλα η τροχαία θα πρέπει να ενημερώσει τα θύματα ή κάθε άλλο δικαιούχο και αυτό θα πρέπει να γίνει με σαφή τρόπο και θα έλεγα να αναπόφευκτα και κατά ανάγκη επιτακτικά στη γλώσσα του συγκεκριμένου ατόμου ότι υπάρχει ένα ε, υπάρχει έννοια της παραγραφής και έχει και κάποια γενική προθεσμία. Αυτά δεν μπορεί να τα εξηγήσει κανείς ε, με ένα φυλάδιο των δύο-τριών σελίδων, αλλά πρέπει να το εξηγήσει τέλο πάντων κάποια στιγμή. Σε ό,τι αφορά τώρα την προθεσμία, Φυσικά και ήταν λογικό να αναζητηθεί μια εναρμόνιση μεταξύ των κρατών μελών. Ε, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αποφυγή μια σειρά από προβλημάτων και συμβάντων, ενώ θα παρέχει και μια προφανή υπηρεσία στον Ευρωπαίο πολίτη. Και αφού αυτή η εναρμόνιση δεν έχει καμία οικονομική επίπτωση, δεν φαίνεται να δημιουργείται πρόβλημα, στα μάτια των θυμάτων. Επομένως, με αυτή την προθεσμία, την αρμοσμένη, τη γενική, λίγη σβήνει το δικαίωμα ε, αποκα... διεκδίκησης, αξίωσης, αποζημίωσης. Θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη μια τέτοια προθεσμία. Τις επιπτώσεις ε, και τις βλάβες που παραμένουν, άρα δεν μπορεί να είναι μικρή αυτή η προθεσμία, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη και το ψυχικό, εγκεφαλικό στοιχείο, ότι δηλαδή πολλές φορές η δήλωση γίνεται πολύ μετά το τροχαίο. Πέντε-έξι ε, χρόνια, δέκα στη Γαλλία, είναι αρκετά μακρύ σωστό, αλλά ένα, μια πενταετία, εξαετία θεωρώ ότι είναι λογική προθεσμία. Διότι έχουμε κάποιες ε, αρνητικές από τις μπορεί να εμφανιστούν πολύ μετά το τροχαίο. και είναι και σημαντικό για να υπάρχει ένα είδος βεβαιότητας για την κοινωνία και για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Τώρα, η ε, Ομοσπονδία μας ε, ενδιαφέρεται ιδιαίτερα και να, να δει τι ε, αποτέλεσμα, τι συνέχεια έχει αυτή η συζήτηση και ακούσαμε και με πολύ ενδιαφέρον τα όσα είπαν οι ασφαλιστές. Ολοκληρώνοντας θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση και σίγουρα χρειάζεται χρόνος αυτό είναι σημαντικό. Η να δεν μπορεί να είναι μικρή. Και νομίζω ότι με ό,τι υπάρχει, με όλε αυτές τι προθεσμίες και διορίσει που υπάρχουν, 5-6 χρόνια όπως είπα, νομίζω ότι είναι εφικτό, είναι ε, δυνατό να επιτύχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι παρότι έχουμε κάποιο χρόνο για ερωτήσεις και απαντήσεις, ε, να το αφήσουμε αυτό για το τέλος ώστε να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Να δώσω τώρα το λόγο στον Δόκτωρ Κρίστιαν Σάλμα ο οποίος θα μας δώσει την ε, οπτική γωνία της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ο Δόκτωρος Σάλμα προέρχεται από την ε, υπηρεσία ερευνών, ε, την Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Υπηρεσία Ερευνών και θα μας εξηγήσει το ρόλο των EADA και αφού ολοκληρώσει θα δούμε ένα μήνυμα σε βίντεο από την δόκτωρα Τζένι Παπέτας. Λοιπόν, έχετε το λόγο αν θέλετε, 10 λεπτά. Ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε, αφού έχουμε μόλις 10 λεπτά, καλύτερα να δούμε το βίντεο που προετοίμασε η Τζένι Παπέτας. Ε, με τα αποτελέσματα της μελέτης που είχε προετοιμαστεί. Μια γενική ενημέρωση, γενικός σκοπός των ευρωπαϊκών τη θέμενης αξίας είναι κατά πόσο να ελέγχει κατά πόσο οι νομοθετικές ε, δράσεις ε, της Ευρώπης σε τομείς όπου δεν υπάρχει ακόμα πολιτική θα δημιουργούσε προστιθέμενη αξία για τους πολίτες και αυτός είναι ο γενικός σκοπός ε, της μελέτης της κυρίας Παπέτας και του κυρίου Μπάνου. Και αν υπάρχουν ερωτήσεις τα μέλη του γύρω σεκρεταρίατα του προσωπικού και εγώ θα μπορέσουμε να τα διαβάσουμε και να λάβετε απαντήσεις Σε Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον τεχνικά είμαστε έτοιμοι να δούμε, να προβάλλουμε το βίντεο. Καλημέρα, θα σας μιλήσω για την αναρμόνιση των περίοδων παραγραφής. Λυπάμαι που δεν μπορώ να βρίσκομαι μέσα σήμερα. Τη μελέτη εξήγαγε ο κύριο Μπόνα και εγώ και εξετάσαμε το κατά πόσο οι κανόνε παραγραφή θα πρέπει να εναρμονιστούν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά αξιώσει που προκύπτουν από διασυνοριακά οδικά ατυχήματα. Εγώ ήρθα στι Βρυξέλλε το Φεβρουάριο για να παρουσιάσω τα ενδιάμεσα ευρήματα τη μελέτη και καλό θα ήταν να επαναλάβουμε ορισμένε από τι παρατηρήσει που έκανα τότε και να παρουσιάσουμε τι τελικέ συστάσει τη έκθεση. Η έκθεση εστιάζεται στις χρονικές προθεσμίες που εφαρμόζονται για την υποβολή μιας αξίωσης. Εάν σε κάποια κράτη-μέλη δεν υπάρχει τέτοια συμμόρφωση με αυτές τις προθεσμίες, τότε χάνεται η δυνατότητα. Αυτή είναι οι κανόνες παραγραφή. Σε άλλα κράτη-μέλη, εάν δεν υπάρχει συμμόρφωση με την προθεσμία, το ίδιο το δικαίωμα διαγράφεται. Και αυτή είναι οι κανόνες παραγραφής. Και στις δύο περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι το ίδιο υπάρχει απώλεια του δικαιώματος ε, υποβολής αξίωσης και έτσι ε, χάνει ο εναγών ε, το δικαίωμα του να έχει πρόσβαση στην δικαιοσύνη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει δυνατότητα υποβολής αξίωσης κατά ενός ασφαλιστικού οργανισμού στο κράτος μέλος όπου διαμένει. Έτσι τα θύματα έχουν ένα οικείο νομικό περιβάλλον και τη δυνατότητα να διεξάγουν τη διαδικασία στη δική τους γλώσσα, σε μια διαδικασία που είναι γνωστή σε αυτούς και στους νομικούς συμβούλους τους. Για το ποιο ε, νομοθεσία πρέπει να εφαρμόζεται, συνήθως εφαρμοστεί η νομοθεσία του τόπου όπου έγινε το ατύχημα. Παρότι δηλαδή πολλοί μπορούν να υποβάλουν την αίτηση αξίωση ε, στη δική του χώρα, πολύ συχνά η νομοθεσία που εφαρμόζεται είναι ξένοι και συνεπώς άγνωστοι. Και εδώ υιοτίθεται το θέμα των κανονών παραγραφής. Όπως είπα το Φεβρουάριο αυτό δημιουργεί διάφορες δυσκολίες για τους ενάγοντες. Firstly, uh, and most Πρώτα απ' όλα και πρωταρχικά, ε, αν οι κανόνες παραγραφής δεν, είναι, δεν έχουν γίνει κατανοητοί, μπορεί να απολεστεί το δικαίωμα αξίωσης. Οι κανόνες ε, παραγραφής είναι περίπλοκοι, αφορούν το συνολικό, τη συνολική χρονικό όριο, το πότε πρέπει να ξεκινά, η χρονική περίοδος, πότε μπορεί να διακοπεί προσωρινά, πώς λειτουργούν οι κανόνες σε σχέση με τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρίες και κατά πόσο το δικαστήριο έχει τη διακριτική ευχαίρεια να αποφασίσει για την εφαρμογή των κανόνων. Κάθε κρατό μέλο έχει διαφορετικού κανόνε για κάθε μία από αυτέ τι πτυχέ και έτσι το νομικό το οποίο είναι διαφορετικό και μοναδικό σε κάθε κράτο μέλο και αυτό απαιτεί εξειδικευμένε γνώσει. Επίση πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι πιο δύσκολη η οργάνωση μια αξίωση από το εξωτερικό σε γενικέ γραμμέ. Χρειάζεται χρόνο, να βρει κάποιος το σωστό εκπρόσωπο ή ασφαλιστή, να συλλέξει στοιχεία για το ατύχημα και να συγκεντρώσει ε, όλα τα παραταγράφα και να τα μεταφράσει. Υπάρχουν παραδείγματα υποθέσεων όπου η έλλειψη γνώσης του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι κανόνες παραγραφής οδήγησε σε απώλεια του δικαιώματος αξίωσης ε, για τον ενάγοντα. Ε, αλλά πέραν αυτού η εφαρμογή ε, ξένων περιόδων δημιουργεί επιπλέον εμπόδια για τους ενάγοντες που προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Η κατάσταση συχνά απαιτεί ε, να, αφιερώσει περισσότερες ώρες ο νομικός σύμβουλος ε, για να ασχοληθεί με το ζήτημα της παραγραφής και αυτό συνεπάγεται επιπλέον δαπάνε. Και επιπλέον δαπάνε υπάρχουν επίσης εάν κληθεί κάποιος εμπειρογνώμων της χώρας του ατυχήματος για να παρέχει συμβουλέ. Αυτά τα εμπόδια είναι αρκετά τακτικά. Αυτά τα επιπλέον εμπόδια αντίκειται στους σκοπούς των κανόνων προστασίας της οδηγίας MID που υποτίθεται ότι διευκολύνει την ελευθερία διακίνηση των ατόμων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Μπόνα και εγώ πιστεύουμε ότι η εναρμόνιση των κανόνων παραγραφής θα έχει σημαντικά πλέον Αυτή η εναρμόνιση θα οδηγούσε σε εφαρμογή κανόνων όσον αφορά δράσεις που προβλέπονται από την Οδηγία Οδικών Ασφαλίσεων, δηλαδή δράσεων ε, αγωγών κατά ασφαλιστών και αγωγών κατά οργανισμών αποζημίωσης για υποθέσεις διασυνοριακής φύσης. Ε, αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με μια τροπολογία της οδηγίας. Η ευθύνη για την ευθύνη των προϊόντων είναι ένα καλό παράδειγμα εναρμόνισης των κανόνων παραγραφής. Στην εκθέση μας λοιπόν συνιστούμε μια ελάχιστη αναρμονή των προτύπων που θα περιλαμβάνει τετραετή συνολική ε, προθεσμία η οποία θα ξεκινάει από την ημερομηνία κατά την οποία ο ενάγων έχει τη γνώση της πλήρους βλάβης που έχει υποστεί καθώς και το εναντί πρέπει να υποβάλουν την αγωγή θα πρέπει να διακόπτεται το χρονικό διάστημα μόλις ε, η αξίωση υποβληθεί σε έναν ασφαλιστή, έναν εκπρόσωπο αξιώσεων ή έναν οργανισμό αποζημίωσης έως ότου απορριφθεί η αξίωση από το εν λόγω μέρος. Ο χρόνος ε, που παραμένει θα πρέπει να λύγει σε όχι λιγότερο από έξι μήνες και δεν θα πρέπει να τρέχει ο χρόνος αυτός ε, έναντι ανηλίκων μέχρι να φτάσουν στην ενηλικίωση ή έναντι ατόμων με αναπηρίες έως ότου παύουν να υφίστανται την κατάσταση τη αναπηρία. Η αναρμόνιση φυσικά δεν θα δημιουργήσει ένα απόλυτα ομοιόμορφο σύστημα παραγραφή σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά οι κανόνε αναρμόνιση που προβλέπουν τα ελάχιστα πρότυπα θα βοηθήσουν να αντιμετωπιστούν τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ανάγοντε, παρέχοντα του μια καλή εικόνα του κατά πόσο ε, έχει νόημα να υποβάλουν την αξία αυτή εναντί ενό ασφαλιστή ή ενό οργανισμού και ε, συμπορφωνούνται και με τι αρχέ τη αναλογικότητα και τη επικουρικότητα. Και επίση θα καθησυχάσουν πολλέ από τι ανησυχίε που εκφράζονται ε, από την ε, τομέα των ασφαλιστικών εταιριών όσον αφορά αυτή την ιδέα τη αναρμόνιση. Μια τροπολογία τη οδηγία θα μπορούσε να βασιστεί στο άρθρο 81 τη Συνθήκη Λειτουργία Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο συγκεκριμένα στο 81.2c που προβλέπει την υιοθέτηση μέτρων με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Παρότι η εναρμόνιση μπορεί να επηρεάσει του κανόνε, οι οποίοι είναι ουσιώδει ορισμένα κράτη-μέλη και διαδικαστική μόνο σε άλλα, το άρθρο 81 δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε περιορισμό όσον αφορά του κανόνε τύπου που μπορούν να εναρμονιστούν. Παρότι η οδηγία για την ευθύνη των προϊόντων έχει διαφορετική νομική βάση, όπω φαίνεται δεν υπήρξαν ιδιαίτερε δυσκολίε για τα κράτη-μέλη να ενσωματώσουν του εναρμονισμένου κανόνε παραγραφή από αυτό το μέτρο. Όσον αφορά την προστιθέμενη αξία της αναρμόνισης, όπως τόνισα το Φεβρουάριο, ο ακριβής υπολογισμός της προστιθέμενης αξίας δεν είναι κάτι εύκολο, διότι δεν υπάρχουν τα απαραίτητα στατιστικά δεδομένα όσον αφορά τον αριθμό ατυχημάτων που λαμβάνουν χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώ καθώς και το πόσο από αυτά τα ατυχημάτα οδηγούν σε αξιώσεις όπου τίθεται το ζήτημα της παραγραφής αλλά έχουμε κάποιες βασικές ε, γενικές ενδείξεις όσον αφορά την πιθανή προσθέμενη αξία σε νομισματικά στοιχεία ε, σε περίπτωση εναρμόνισης. Τα νούμερα που υπάρχουν στην έκθεση λαμβάνουν υπόψη ατυχήματα με σωματική βλάβη ή θάνατο, αλλά και ατυχήματα με μόνο υλικέ ζημιέ. Τα ατυχήματα με μόνο υλικέ ζημιέ ε, θα είναι πιθανότατα ε, το μεγαλύτερο ποσοστό ατυχημάτων γενικότερα και πολύ συχνά δεν δηλώνονται. Η βελτίωση τη πρόσβαση στη δικαιοσύνη για αυτά τα θύματα είναι σημαντική. Συνήθω εστιαζόμαστε σε άτομα που υπέστησαν σωματική βλάβη και που σαφώς χρειάζονται αποζημίωση για τη βλάβη αυτή. Ωστόσο η χρήση των ε, αυτοκινήτων ε, έχει πολύ σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές ε, εφαρμογές και η υποστήριξη προς όσους χρειάζονται απλά επισκευή του αυτοκινήτου τους, η αντικατάσταση του αυτοκινήτου τους είναι επίση σημαντική. Ε, τα στοιχεία δείχνουν ότι όσοι χάσουν το δικαίωμα αξίωση χάνουν κατά μέσο όρο 16.000 ευρώ για προσωπικές βλάβες και 2.000 περίπου για ε, καθαρά υλικέ βλάβες. Και αυτό φυσικά δεν αντικατοπτρίζει τις τραγικές ε, συνέπειες που έχει μια καταστροφική σωματική βλάβη σε περίπτωση απώλειας του δικαιώματο. Βασί των αναλύσεων μα περίπου 250.000 άνθρωποι έχουν αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα παραγραφής ε, ετησίως. Το μέσο επιπλέον νομικό κόστος που σχετίζεται με τα ζητήματα παραγραφής ε, υπολογίζεται στα 600 περίπου ευρώ αναξίωση και το κόστος ε, της αναζήτησης συμβουλευτικής υποστήριξης από υπερογνώμονες είναι περίπου 300. Συνολικά λοιπόν η εναρμόνιση θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξοικονόμηση 300 εκατομμυρίων ετησίω. Το νούμερο αυτό δεν λαμβάνει υπόψη τις δαπάνες που σχετίζονται με επιπλέον δικαστικά έξοδα ή έξοδα μετάφρασης γιατί δεν έχουμε στοιχεία για αυτά τα ζητήματα αυτή τη στιγμή. Αλλά όπως φαντάζεστε η εξοδα μεταφραση γιατι προσθέμενη αξία θα είναι ακόμα υψηλότερη. Η πραγματικη προσθεμενη κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και ιδιαίτερα περίπλοκη δημιουργώντας τεράστια βεβαιότητα για τα μέρη ε, που θα ήθελαν να υποβάλουν κάποια αξίωση σε περίπτωση διασυνοριακού οδικού ατυχήματος για λόγους παραγραφής. Η εναρμόνιση των κανόνων παραγραφής θα μπορούσε να ε, παράσχει ε, πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θύματα ατυχημάτων και να βοηθήσει την ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανάλυση μας δείχνει ότι πολλοί άνθρωποι επηρεάζονται από αυτό το ζήτημα ετησίω και ότι προβλέπονται σημαντικέ εξοικονομήσει σε περίπτωση εναρμόνισης. Ευπίζουμε τα πορίσματα της μελέτης μας να σας φανούν χρήσιμα και το Κοινοβούλιο να λάβει δράση επί του ζητήματος και να κινηθεί το όσο το δυνατόν ταχύτερα. Εδώ ολοκληρώνεται η παρουσίασή μου. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Okay. We Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση αυτή. Μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε με την προοπτική της Κομισιόν. Ε? Ελπίζω ο κύριος Γκέορκ Χάιμπαχ να είναι εδώ. Είναι? είναι ανώτερος ε, νομοθετικός ε, αξιωματούχος ε, στη μονάδα πολιτικής αστικής δικαιοσύνης σε διεύθυνση Α, δικαιοσύνη, 10 λεπτά και εσείς παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως γνωρίζετε, Σύμφωνα με τα 4 και 15H ε, του κανονισμού Ρώμη 2, οι εφαρμοστές προθεσμίες ε, για την υποβολή αξιώσεων ε, ορίζονται καταρχήν από το δίκαιο της χώρας όπου συνέβη το τροχαίο. Αυτοί οι κανόνες λοιπόν, από τον κανονισμό της Ρώμης 2 έχουν αυξήσει την ασφάλεια δικαίου σήμερα. Ένας κανόνας ορίζει τις προθεσμίες. Ο κανόνας, ο νόμος αυτός ισχύει οπουδήποτε γύρεται η αγωγή σε οποιοδήποτε κράτος μας. Φυσικά υπάρχουν διαφορές μεταξύ εθνικού αστικού δικαίου, περιόδων ε, περιορισμού ε, παραμένουν αυτές οι δυσκολίες και αυτό δημιουργεί πρακτικά προβλήματα, ιδίω γιατί πρέπει κανείς να γνωρίζει το αλλοδαπό δίκαιο και κάποιες φορές αυτό δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες που ενδέχεται να έχουν οι πολίτες, ιδίω αν το εφαρμοστέο δίκαιο είναι λιγότερο ευνοϊκό από το δίκαιο που ισχύει στη δική τους χώρα. Ωστόσο, το βασικό αποτέλεσμα ε, της μελέτης και των δημόσιων διαβουλεύσεων που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών για το ισχύον δίκαιο. Και αυτό το κάναμε. Είχαμε λοιπόν ε, καταρχάς μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ξεκίνησε το 2008 η μελέτη της Κομισιόν ε, που μελέτησε διάφορες επιλογές για να βελτιωθεί η κατάσταση. Και με βάση αυτή τη ε, μελέτη έγιναν δύο διαβουλεύσεις, η μία το 2009 και η δεύτερη το 2012. Το αναφέραμε προηγουμένως αυτό. Ποια ήταν η ανταπόκριση. Οι απαντήσεις συνήθως ε, αντικατέτριζαν ε, τα συμφέροντα των κλάδων. Οι ασφαλιστές παραδείγματος χάρη βλέπουν κάποια προβλήματα ε, με μια μικρή προθεσμία. Να είναι ελάχιστα ή να μην μπορούν να μετρηθούν. Άρα δεν θεωρώ ότι χρειάζεται να αναλυφθεί δράση. Τα θύματα, κατά την άποψή τους, ε, αξιοποιούν την νομική συμβουλή και αντιδρούν ε, εγκαίρω. Προστασία θυμάτων τώρα. Οι οργανισμοί, οι δικηγόροι περάσπιση. έδωσαν παραδείγματα για τις διαφορές μεταξύ των εθνικών περιόδων. Ότι δηλαδή υπήρξαν περιπτώσει που δεν ε, πήραν την αποζημίωση στα θύματα. Οι ασφαλιστές είναι λοιπόν κατά μιας πιθανής εναρμόνισης, ενώ άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς που εστιάζουν κυρίως ε, στα θύματα είναι πιο ανοιχτοί σε αυτή την ιδέα. Πάντω υπάρχει συμφωνία ότι χρήζει βελτίωση ανταλλαγή πληροφοριών. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να υπάρξουν εθνικά δελτία αναλυτικά που θα περιγράφουν τι προθεσμίε που ισχύουν σε κάθε κράτο μέλο. Σε συνέχεια της διαβούλευσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το παραδοσιακό ε, δίκτυο που έχει για τα αστικά και ποινικά θέματα, δημοσιοποίησε ε, στην πύλη του, της ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ δικαιοσύνης κάποια δελτία. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τα δούμε. Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε το σύνδεσμο, την ιστοσελίδα. Ναι, εδώ ακριβώς. Βλέπετε λοιπόν εδώ το link στη πύλη, τη διαδικτυακή πύλη, η Justice, και εκεί μπορείτε να δείτε αυτά τα δελτία. Αυτό είναι σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της κατάστασης, δηλαδή δίνουν περισσότερες πληροφορίες και μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην επίτευξη του στόχου να αποφύγουμε ανεπιθύμητες ε, επιπτώσεις ε, για τα θύματα των διασυνοριακών τροχαίων. Επειδή διαφέρουν το συστικό δίκαιο της μιας χώρας από την άλλη, σε ό,τι αφορά τους περιορισμούς και τις προθεσμίες ότι η δράση αναλυφθεί για την εναρμόνιση αυτών των ε, περιόδων θα πρέπει να σεβαστεί την αρχή της επικουρικότητας και να δοκιμαστεί. Οι προθεσμίες ε, δεν είναι κάτι απομονωμένο, αλλά εντάσσεται στις γενικότερες ε, διατάξεις του δικαίου και των κωδίκων αστικής δικονομίας, πολιτικής δικονομίας. Τώρα μελετούμε τα τελικά πορίσματα στην Κομισιόν. Σας παρουσίασα τα βασικά. Ποιο είναι το συμπέρασμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση, ιδίω υπό το πρίσμα των πληροφοριών και των δράσεων που έχουν μέχρι τώρα αναλυφθεί και βέβαια υπό το φως πληροφοριών για προβλήματα που θα απαιτήσουν περαιτέρω δράση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς ήσταν ο τελευταίος ομιλητής ε, σε αυτή την ακρόαση. Άρα δηλαδή έχουμε τώρα χρόνο για ερωτήσεις και ελπίζω να δοθούν και απαντήσεις. Και απευθύνομαι στα μέλη. Δεν ξέρω, θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Ο κ. Λεμποχατών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Καταρχάς, να ευχαριστήσω όλους ε, τους ομιλητές που ήρθαν και εξέφρασαν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες απόψεις και συγκεκριμένα τον κύριο Βάντεργκεμ, το οποίου σκοτώνω και εγώ το όνομα δυστυχώς. Ε, ε, αναγνωρίζω το γεγονός ότι μίλησε γαλλικά, παρόλο που είναι Ολλανδός, βλέπω ένα καλό σημάδι για τη συνέχιση των εργασιών μας. Ο κύριος ε, Ζανμέρκ μίλησε ε, αγγλικά. Ευτυχώς έχουμε τους εξαιρετικούς αυτούς τους διερμηνείς που μας επιτρέπουν να μιλάμε την εθνική μας γλώσσα. Εγώ συνήθως δεν μιλώ ε, αγγλικά. Εχθές όμως στην Επιτροπή Ελευθεριών δεν υπήρχε διερμηνέας. Είναι σκάνδαλο. Και αναγκάστηκα να μιλήσω αγγλικά. Φτάνω στην ουσία τώρα. Το θέμα σήμερα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και σοβαρό γιατί έχει να κάνει με τις προθεσμίες παραγραφής ε, όταν μιλάμε για προσφυγές μετά από τροχαία ατυχήματα και αυτό ε, που είναι σημαντικό εδώ είναι ότι έχουμε δύο ε, στρατόπεδα, δύο λύσεις για να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ποικιλομορφίας, της προθεσμίας αυτές στα κράτη-μέλη. Ε, έχουμε πρώτα το στρατόπεδο της εναρμόνισης, να κάνουμε κανόνες νομικούς που θα εναρμονίσουν τα εθνικά δίκαια. Νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι οι ομιλητές που ήρθαν σήμερα εδώ υπερασπίζονται αυτή την θέση εκτός από τον κύριο Ζανμάρ. Και ε, το δεύτερο στρατόπεδο που αυτός εκπροσωπεί είναι αυτό των ασφαλιών που επιλέγει μια άλλη λύση, μια καλύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες. Να εξηγούμε δηλαδή στα θύματα ότι οι κανόνες δικαίου που ισχύουν σε άλλες χώρες δεν είναι οι ίδιες, οι ίδιοι με, στη χώρα τους, άρα μπορεί να διαφέρουν και οι προθεσμίες παραγραφής. Εγώ, δεν με ξέρουν ίσως οι ομιλητές, αλλά εγώ να πω ότι θα επέλεγα τη λύση της καλύτερης πρόσβασης στις πληροφορίες παρά την εναρμόνιση. Γιατί θα σας το εξηγήσω σύντομα και θα ολοκληρώσουμε μια ερώτηση. Πρώτον, διότι είναι ε, πολλά τα προβλήματα που σχετίζονται με την ποικιλομορφία, δεν είναι πολλά αυτά τα προβλήματα που σχετίζονται με την ποικιλομορφία ε, στις προθεσμίες. Ο κύριος Ζανμάρ που εκπροσωπεί τις ασφαλιστικές εταιρείες συμφωνεί και υπογραμμίζει ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν μέσω καλύτερης πληροφόρησης. Ο τρίτος λόγος είναι μία αντίρρηση σε κάτι που μας υπόθηκε στο βίντεο. Ε, λέγεται ότι η εναρμόνιση θα μας βοηθήσει να εξοικονομήσουμε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σύμφωνα με τους υπολογισμούς και κάτι τέτοια. Εγώ δεν έχω πιστεί να μην μας τα πουλάνε αυτά κάθε φορά, να μην μας πουλάνε την εναρμόνιση ε, λέγοντας ότι θα ξεκονομήσουμε χρήματα, γιατί στην πραγματικότητα δεν το ξέρουμε. Δεν ισχύει το επιχείρημα. Και τέλος, το βασικό μου επιχείρημα είναι η επικουρικότητα φυσικά είναι, ε, είμαι πάντοτε ε, υπέρ της επικορικότητας η οποία ε, συνεχώς αναφέρεται αλλά ξεχνάμε την ουσία της. Σήμερα αυτή που είναι υπέρ της εναρμόνισης ανέφεραν την επικορικότητα. Αυτό είναι περίεργο γιατί για μένα το αντίθετο πρέπει να γίνεται, να την αναφέρουμε όταν μιλάμε για τις εθνικές ιδιαιτερότητες που πρέπει να αφαιθούν να υπάρχουν και όχι για εναρμόνιση. Από εδώ και πέρα φαίνεται ότι γίνεται και αυτό. Για να ολοκληρώσω θα αναφέρω μία φράση του κυρίου Έμπακ που είπε ότι πρέπει να γνωρίζουμε τα ξένα δίκαια όταν είμαστε θύματα ενός τροχαίου ατυχήματος. Με τρόμαξε αυτό, όντως είναι ένα μειονέκτημα, αλλά με μία ε, με ένα τέτοιο επιχείρημα θα έπρεπε να καταργήσουμε κάθε είδους εθνική νομοθεσία, γιατί δημιουργεί προβλήματα στους ανθρώπους. Όμως ε, τα κράτη έχουν τις ιδιαιτερότητές τους ε, που τις θέλουν και εγώ τις σέβομαι στο μέγιστο και νομίζω ότι στα τροχέα η καλύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες θα έφτανε για να λύσουμε το πρόβλημα που ενδεχομένως προκύψει κάποια στιγμή. Να φτάσω λοιπόν στην ερώτησή μου. Τι μπορείτε να μου πείτε για να με πείσετε, αφού είστε οι περισσότεροι υπέρ της εναρμόνισης, ποιο είναι το βασικό επιχείρημα που θα μου δίνατε για να με πείσετε ότι η εναρμόνιση εδώ επιβάλλεται σε σχέση με την βελτίωση της πρόσβασης της πληροφορίας. Ευχαριστούμε κύριε Λεμπρετών, ο κύριος Αλέφ. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστούμε τους συμπρογνώμονες για τις λεπτομέρειες πληροφορίες που μας παρουσίασαν. Όπως φαίνεται, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, υπάρχουν σημαντικές διαφορές ε, και αποστάσεις όσον αφορά τις προθεσμίες παραγραφής. Σε ορισμένα κράτη-μέλη, οι προθεσμίες αυτές ε, εξαρτώνται από το αν πράξη ε, ε, αποτελεί παραβίαση ή από τον τύπο του ατυχήματο. Και βλέπουμε ότι αυτέ οι διαφορέ μπορούν να οδηγήσουν σε ανεπιθύμητε συνέπειε για τα θύματα των ατυχημάτων και να δημιουργήσουν επιπλέον ε, προσκόμματα για τα θέματα. Υπάρχει ένας πραγματικός κίνδυνος διασυναριακών ατυχημάτων για τα θύματα όταν υποβαλούν αγωγή αποζημίωσης. Λόγω αυτών των διαφορών των ε, νομικών αποστάσεων σε θέματα αποζημίωσης και σε θέμα εφαρμοστέου δικαίου Λόγω όλων αυτών λοιπόν ε, η έκβαση των ε, υποθέσεων ε, επηρεάζεται ιδιαίτερο σε ορισμένες ε, περιπτώσεις. Εάν το κράτος ε, διαμονής του θύματος και του υπευθύνου είναι το ίδιο, εφαρμόζεται αυτό εν λόγω δίκαιο. Σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης, το κράτος όπου έχει εγγραφεί το αυτοκίνητο και το συγκεκριμένο δίκαιο έχουν εφαρμογή. Πώς μπορούμε να καλύψουμε αυτές τις διαφορές μεταξύ της Χάγης και του κανονισμού ώστε να εφαρμοστούν όλα αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ έχω μια ερώτηση. Η δική μας Επιτροπή έχει συστήσει μια ομάδα εργασίας για τη ρομποτική και για αντιοντολογικά θέματα της οποίας προεδρεύει η Αντελβό και στο πλαίσιο αυτής της ε, ομάδας ε, εργασίας έχουν θέσει θέματα ευθύνης οδηγού. Ε, έτσι λοιπόν η υπηρεσία ΣΥ έχει δημοσιεύσει μία μελέτη για τα τροχαία ατυχήματα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα ατυχήματα που μπορούν να προκύψουν από οχήματα χωρίς οδηγό. Πιστεύετε ότι μπορούν να προκύψουν και εκεί ε, θέματα παραγραφής όταν προκαλούνται τροχαία ατυχήματα από αυτοκινούμενα οχήματα. Και τι πιστεύετε και για την περίπτωση θανάτου. Υπήρξε ένας θάνατος που προκλήθηκε από ένα όχημα χωρίς οδηγό. Αυτόματα. Οχήματα. Δεν ξέρω. Θέλετε να τοποθετηθείτε από αυτό που ακούσατε. Αν ναι, παρακαλώ να λάβετε το λόγο. Πρόεδρε, εγώ να πάρω πρώτος το λόγο γιατί μίλησα και πρώτος. Είμαι ο Φίλιπ Μίντ. Όσον αφορά λοιπόν στο να απαντήσουμε στο πρώτο ερώτημα και να πείσουμε τον ερωτώντα ξαρτάται από το ποιο είναι, το σημείο κίνησή σας. Όπως και στο Brexit οι άνθρωποι μερικοί είναι μονομανείς, είναι ιδεολειπτικοί, δεν πρόκειται να πιστούν από επιχειρήματα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ε, ότι βασιζόμαστε στην καλύτερη ενημέρωση. Θα αναφέρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα γιατί εξακολουθούμε να είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η περίοδος ε, παραγραφής στην Ισπανία είναι ένας χρόνος και εκεί υπάρχουν ε, σοβαρά ατυχήματα, προκαλείται ζημιά ψυχιατρικής φύσεως και κατά το πρώτο έτος δεν είναι σε θέση να καταλήξουν στο κατά πόσον θα κατατεθεί αγωγή. Όχι, γιατί σας είπα, υπάρχουν τα μεγάλα ψυχιατρικά τραύματα. Αποκτούν τις καλύτερες πληροφορίες που μπορούν από το, την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί αναφέρεται ότι η αγωγή πρέπει να κατατεθεί εντός του έτους. Και δεν έχουν συνειδητοποίηση ότι η ημερομηνία είναι η ημερομηνία σταθεροποίησης date of stabilization τι σημαίνει αυτό για ε, έναν Εγγλέζο αυτό δεν υφίσταται ο, ε, ο χρόνος τρέχει από την ημερομηνία που λαμβάνει η χώρα το τροχαίο τύχημα date of action επίσης ε, ε, ούτε ξέρουν και πώς λειτουργεί όλο αυτό το ποινικό σύστημα στην Ισπανία. Άρα δηλαδή σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος ένας άνθρωπος που είναι καλά πληροφορημένος παρόλα αυτά να μην πάει στο δικηγόρο γιατί μπορεί να πει είδα την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μου λέει ότι υπάρχει περιτόριο μόνο ενός έτους, ο χρόνος έχει περάσει, ε, τέλειος ιστορία γιατί ε, να δαπανώ τα χρήματά μου σε δικηγόρους έτσι κι αλλιώς έχασα την προθεσμία. Αυτή μπορεί να είναι η άποψη του ε, ενδιαφερόμενου. Άρα δηλαδή υπάρχει μια άποψη ότι τα ξέρουν όλοι οι δικηγόροι και κανείς άλλος. Αυτοί είναι και οι καλύτεροι πελάτες των δικηγόρων. Μα κάποιες γνώσεις, λίγες νομικές γνώσεις, ε, βεβαίως και δεν μπορούν να σε βοηθήσουν για να επιτύχεις το στόχο Το θέμα ότι όλο αυτό είναι τόσο περίπλοκο υπάρχει και δεν μπορεί να εναρμονιστεί. Αυτή είναι η απάντηση. Αν τα πράγματα είναι τόσο περίπλοκα που δεν μπορούν να εναρμονιστούν, ε, και δεν μπορούν να λυθούν τα προβλήματα με τις πύλες και τα ενημερωτικά φυλάδια. Το θέμα είναι πάρα πολύ δύσκολο και αν δεν υπάρχουν γενικές ε, περιόδους απόσβεσης, αλλά υπάρχει κάποια ειδική εναρμόνιση σε σχέση μόνο με ειδικέ ε, οδηγίες, γιατί αυτά άκουσα μέχρι τώρα και ε, από ό,τι κατάλαβα η Jennifer Peepers τα είπε αυτά. Υπάρχει λοιπόν ένα δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών και είναι ευρωπαϊκή απόφαση που πρέπει να ληφθεί για να εναρμονιστούν οι περίοδοι εναρμόνισης με βάση αυτά που ισχύουν κάτω από το πρίσμα της κοινή αγοράς. Εγώ λοιπόν θέλω να πω ότι η επικουρικότητα, αν θέλετε τη σωστή δράση, τότε αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν και οι σωστοί κανόνες που θα είναι ο συγκερασμός επικουρικότητας και λογικής και να υπάρχει και κάποια αναλογικότητα. Εν ολίγης, αυτά είχα να πω. Τώρα δεν ξέρω αν σας έπεισα, αλλά εγώ αυτά είχα να πω. Όσον αφορά στις διαφορές ανάμεσα αποφάσεις του Δικαστηρίου της Χάγης και της απόφασης Ρώμη 2, πράγματι οι διαφορές είναι πολύ μεγάλες, αλλά ο κανονισμός Ρώμη 2 και ο κανονισμός της Χάγης δεν διευκολύνουν την κατάσταση. Ε, ο κανονισμός ε, Ρώμη 2 έχει περιπλέξει τα πράγματα. Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις χώρες που έχουν προσυπογράψει ή έχουν υιοθετήσει αυτόν τον κανονισμό και άλλες που δεν τον έχουν δεχτεί, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι πράγματι όλο αυτό είναι πάρα πολύ περίπλοκο. Φταίει και ο κανονισμός Ρώμη 2 και εγώ πιστεύω ότι αν θέλει να τα πλουστεύσει κανείς κάπως τα πράγματα, τότε θα πρέπει να πλουστεύσει όλα αυτά που αναφέρονται στο κανονισμό Ρώμη 2. Όσον αφορά τη ρομποτική, να πω κάτι που ίσως να μην είναι απόλυτα αυτονόητο, αλλά όπως και στη Γαλλία δεν υπάρχει ευθύνη για επαιτιότητα υπάρχει και αστική ευθύνη που προκύπτει λόγω ατυχήματος. Θα μπορούσε κανείς να εθετήσει ένα παρεμφερή κανόνα. Και ε, υπάρχει και ένα καθεστώς που ίσως να μην το κρίνατε σημαντικό, όμως ε, θα μπορούσε να προσφέρει τη λύση. Ας πούμε ο χώρος. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες ε, όσον, μάλλον το διάστημα το διάστημα, εκεί θα μπορούσε να ζητηθεί η λύση, με συγχωρείτε όχι χώρος, διάστημα. Υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς για τα διαστημόπλια και υπάρχει και η σύμβαση των Αθηνών για την Ναυτιλία. Για μένα η ρομποτική είναι άλλος ένας ε, συγκεκριμένος τομέας, ε, εντάσσεται σε θέματα μεταφορών και Συγκρίνοντας το τι ισχύει στις ΗΠΑ, έχουμε προχωρήσει. Και αυτό που λέμε θα μπορούσε ίσως να υιοθετηθεί σε διεθνές επίπεδο. Ευχαριστώ κύριε Ζαν Μάρκ. Να σας ζητήσω να είστε σύντομοι γιατί ήδη χρησιμοποιούμε τον ελεύθερο χρόνο των διερμηνέων μας. Λάβετε το υπόψη παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ. Θα συνεχίσω στα αγγλικά γιατί είναι η γλώσσα εργασίας ε, στην Ένωσή μου. Θα ξεκινήσω με την τελευταία ερώτηση για τη ρομποτική, γιατί κατανοείται ότι η συζήτηση για τα ε, οχήματα χωρίς ε, οδηγό είναι ένα θέμα που συζητούμε πάρα πολύ στην Αντίστοιχη Επιτροπή στην Κομισιόν. Συζητάμε τα ρυθμιστικά θέματα, το θέμα της αστικής ευθύνης, κατά πόσο ε, θα ισχύει όταν έχουμε ε, περισσότερα τέτοια αυτοκίνητα αυτόματα στο δρόμο και ε, πλήρως αυτοματοποιημένη οδήγηση, πόσο θα επηρεαστεί η αστική ευθύνη. Η οδηγία για την ασφάλεια των μηχανοκίνητων οχημάτων θα συνεχίσει να αποτελεί καλό πλαίσιο για την οργάνωση των αποζημιώσεων. Γι' αυτό δεν θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη να ακολουθήσουμε την επιλογή της ε, οδηγίας για την ευθύνη για τα προϊόντα. Νομίζω λοιπόν ότι ε, θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα ε, για τα αυτοματοποιημένα αυτοκίνητα, κατά πόσο θα επηρεάσουν τους κανόνες, ειδικά για την παραγραφή, δεν έχει συζητηθεί αρκετά. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι ίσως τελικά να διευκολυνθεί η κατάσταση για να έχουμε καλύτερη αντιμετώπιση των αξιώσεων με αυτόν τον τρόπο, ε, γιατί ε, υπάρχει ένα μια βασική προϋπόθεση να έχουν ε, όλοι πρόσβαση στα δεδομένα του οχήματος ε, για να μπορεί κανείς να κρίνει μια υπόθεση. Οπότε ε, έτσι θα λυθεί το θέμα πιστεύω και πρέπει να το εξετάσουμε. Όσον αφορά τα ερωτήματα για την εναρμόνιση των περιόδων παραγραφής, θα επαναλάβω την άποψη ότι για μας θα ήταν δύσκολο αυτό το εγχείρημα. Να πω ότι πολλοί ομιλητές αναφέρθηκαν σε δυσκολίες που δεν σχετίζονται απαραίτητα με το γεγονός που είναι ότι είναι διαφορετικοί οι κανόνες, αλλά το ότι είναι περίπλοκες οι διαδικασίες στα κράτη-μέλη. Αυτό δεν θα το αντιμετωπίσουμε με την εναρμόνιση των κανόνων για την παραγραφή ή την αποσβεστική προθεσμία. Οπότε με την ε, αντιμετώπιση των προβλημάτων στον τομέα της πληροφόρησης θα έχουμε μια βελτίωση. Αυτά είχα να πω για να ξεκαθαρίσω τις απόψεις μας για αυτές τις δύο πιθανές προσεγγίσεις. Σύντομα, κύριε Λεμπρετών, θα απαντούσα και με ερώτηση. Γιατί να μην εναρμονίσουμε. Γιατί ε, εντάξει, καταλαβαίνω ότι καθένας μπορεί να θέλει να μείνει πιστός στο εθνικό του σύστημα, για, το καταλαβαίνω και ως παλιός ε, δικηγόρος και νομικός. Δεν ε, έχω κάτι να πω εναντίον αυτού, όμως μιλάμε για κοινέ αρχές που θέλουμε να υπερασπιστούμε και ένα θέμα πρακτικό. Είναι απλά, απλώς πρακτικό θέμα, αλλά θα έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις, ε, καταστροφικές τα λέγαμε, αν ε, δεν ε, βελτιώσουμε την κατάσταση στο θέμα της παραγραφής. Η, αυτή η παραγραφή που διαρκεί μεγάλο διάστημα και αντιμετωπίζει τα προβλήματα όλων των θυμάτων ας πούμε με 10 ετή θα ήταν το ιδανικό, αλλά και με 5-6 χρόνια θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα χωρίς να πειράξουμε τα εθνικά συστήματα. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος που θέλει να μιλήσει. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος, οπότε να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές μας, συμπεριλαμβανομένης και της κυρίας Παπέτας που ήταν εδώ ψηφιακά. Να ευχαριστήσω και τους διερμηνείς που μας χάρισαν λίγο παραπάνω χρόνο. Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεισφορά σας.